Αγαπητοί συνάδελφοι, καλημέρα. Σας καλωσορίζω θερμά στη συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Σήμερα το πρωί έχουμε πάρα πολλές ψηφοφορίες στην ημερήσια διάταξη. Αλλά καταρχήν θα ακολουθήσουμε τη σειρά των θεμάτων όπως αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη. Καταρχήν η έγκριση της ημερησίας διάταξης όπου έχω να κάνω τρεις παρατηρήσεις. Η κυρία Κριστίνα ε, Κορτίνες στο σημείο ο 11 μας ζήτησε να, να παρουσιαστεί ε, μάλλον το, το σημείο 9 να, να ε, έρθει πιο γρήγορα διότι πρέπει να φύγει μετά και πριν από τις implementing powers. Όσον αφορά το αυτό 8 ε, ανακοίνωτη της Επιτροπής μια κοινοτική προσέγγιση για την πρόληψη φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών θα χρειαστεί να αναβληθεί γιατί ίσως θα πρέπει να περιλάβουμε και την ε, ε, τη στάχτη του ηφαιστείου της Ισλανδίας και ως εκ τούτου θα πάει λίγο πιο μετά. Επίσης ε, έχουμε ε, μία αντιπροσωπεία ε, η οποία είχε πάει στην Ισλανδία και αυτό πρέπει να το συζητήσουμε όταν θα έρθει και ο πρόεδρος δηλαδή μετά το σημείο 17 αλλά πριν του σημείου 18 αυτή θα είναι η μερίσια διάταξη της συνεδριάσεως εάν δεν έχετε αντίρρηση. Έχουμε ε, ερμηνεία σε όλες τις γλώσσες εκτός εστονικά και λετονικά και στο τρίτο θέμα της ημερησίας διατάξεως ε, βλέπετε ότι ε, η έκθεση Florence θα ψηφιστεί 22 Ιουνίου και η έκθεση Λάγγεν στις 24 ε, Ιουλίου. Η, κυρία Λούκας ε, είναι η ε, πρώτη, η πρώτη πράσινη βουλευτήνα η οποία εξελέγει εις το Βρετανικό Κοινοβούλιο ε, είναι κάτι το οποίο σημειώνουμε, τις ευχόμαστε κάθε ε, επιτυχία. Η έκθεση Τίμπερ θα αναλυφθεί από τον Τσάτου Χάση. Ε, θα παραμείνει δηλαδή στους πρασίνους, αλλά θα το αναλάβει κάποιος συναδελφός της. Επίσης, η Γενική Γραμματεία ε, ε, ονόμασε μία νέα υπεύθυνη για το κλίμα την κυρία Χριστίνα Φιγκέρα στην οποία ευχόμαστε καλή επιτυχία για να παρακολουθήσει τα θέματα αυτά και τις διαπραγματεύσεις οι οποίες μετά την Κοπενχάγη θα εξελιχθούν για την προετοιμασία του Καλκούν. Ε, στο παρελθόν ε, είχε συμμετάσχει σε μία διαπραγμάτευση για την Κοσταρίκα. Ήταν και στο εκτελεστικό γραφείο των λατινοαμερικανικών χωρών ε, άρα έχει μία συγκεκριμένη γενική ιδέα για την κατάσταση του κλίματος. Έχω συντάξει μία επιστολή ε, για την ε, ε, κυρία Φιγκέρας και θέλω να ευχαριστήσω και τον αποχωρήσαντα γενικό γραμματέα ο οποίος πάντοτε μας βοήθησε και έκανε εξαιρετική εργασία. Θα ήθελα να σας πω σχετικά με την ανακοίνωση της προηγούμενης εβδομάδος για την ανάλυση των εναλλακτικών λύσεων ότι πρέπει να ξεπεράσουμε το 20% είναι κάτι το οποίο θα μας θα μας ε, ε, απασχολήσει ε, διότι βλέπω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είχε το θάρρος να προχωρήσει πέραν του 20% και εμείς πρέπει να παίξουμε ένα βασικό ρόλο σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διότι θα πρέπει και την επόμενη εβδομάδα να είμαστε δραστήριοι στο θέμα αυτό. βλέπετε ότι λάμπει ο ήλιος Βλέπετε όμως ότι εμένα θα μου άρεσε, αλλά για την ψηφοφορία κατεβάζουμε τα ρολά. Τώρα, ανακοίνωση της Επιτροπής για το ε, χάρτη πορείας για το χακούν. Είναι κάτι το οποίο θα συζητήσουμε και θα ήθελα να σας πω εν ευθέτω χρόνο. Και θα ήθελα επίσης να σας πω ότι την 5η 10 Ιουνίου από τις 9 και 15 ε, μέχρι τις 12 και 30 θα συζητήσουμε για την στρατηγική της ε, Ευρωπαϊκής Ενώσεως διότι ήταν μια εποχή όπου δεν υπήρχε η δυνατότητα να ασχοληθεί επαρκώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και γι' αυτό είχε διατυπωθεί η επιθυμία να οργανώσει η Επιτροπή Περιβάλλοντος ένα workshop μαζί με όλους τους ενδιαφερόμενους και τους ειδικούς. Άρα στις 18 Ιουνίου είσαστε όλοι προσκεκλημένοι ε, για να συμμετάσχει σε αυτό το συμπόλιο για την ε, αηφορία και ε, επίσης ε, ε, η κυρία Λεπάζ έχει ζητήσει από κάποιον φωτογράφο να έρθει να πάρει φωτογραφίες. Ε, επίσης, ε, όπως σας είπα, το θέμα 8 θα μετατεθεί για την επόμενη συνεδρίαση και τώρα ερχόμαστε στο τέταρτο θέμα, απολογισμό της επίσκεψης αντιπροσωπείας ΕΜΒΗ στην Ισπανία 22-24 Μαρτίου 2010 δηλαδή αρκετά αργά αλλά λόγω της Κοπενχάγης το Δεκέμβριο δεν είχαμε την ευκαιρία να μεταβούμε στην Ισπανία γι' αυτό και το μεταθέσαμε στο Μάρτιο όπου κάναμε πολλές συζητήσεις για την προστασία του κλίματος με τους ειδικούς του περιβάλλοντος ε, διότι θέλαμε να βολιδοσκοπήσουμε τις ε, ε, φιλοδοξίες της Ισπανικής Προεδρίας Προεδρίας να κρατήσει το θέμα αυτό στο επίκεντρο και επίσης στις 23 Μαρτίου στη Μαδρίτη υπήρχε μία παγκόσμια διάσκεψη ε, επί αυτού του θέματος όπου διάφοροι ε, συμμετέχοντες της επιτοπής ε, παρουσιάστηκαν, συμμετείχαν εις την αντιπροσωπεία πήγαν μετέβησαν στο κέντρο ο μεταμοσχεύσεως οργάνων της Ισπανίας που ηγείται στον τομέα αυτό και ε, ε, ελπίζουμε ότι και οι άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσης θα μπορέσουν ε, να φτάσουν το ίδιο υψηλό επίπεδο το οποίο παρουσιάζει η Ισπανία στο θέμα αυτό αυτή τη στιγμή. Είχαμε επίσης επαφές με τους εκπροσώπους του Κοινοβουλίου και της Γερουσίας με τους εκπροσώπους της Επιτροπής μας και εδώ η, ε, υπήρχε ιδιαίτερη, ε, ιδιαίτερη συμμετοχή για το θέμα της σημάνσεως των τροφίμων ε, όσον αφορά τις συσκευασίες. Ήταν ένα σοβαρό θέμα όπως άλλωστε και τα απόβλητα διότι τα απόβλητα είναι ένα σοβαρό πρόβλημα στην Ισπανία δηλαδή πώς θα απομακρύνονται τα πόβλητα. Ε, αύριο το πρωί έχουμε μία συνεδρίαση με τις ισπανικές μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Ε, αυτό είναι κάτι το οποίο έχει προετοιμαστεί πολύ σωστά ε, και όταν ήμασταν στην Ισπανία μας μίλησαν για τα νέα προγράμματα κατασκευής αυτοκινητοδρόμων και σιδηροδρόμων διότι προβλέπεται ε, μία ε, με σιδηροδρομική γραμμή από το Λέδο ε, μέχρι τις ακτές μέσω μιας περιοχής η οποία είναι ε, χαρακτηρισμένη Νατούρα και πρέπει να ελεγχθεί εάν θα γίνουν σεβαστές οι προδιαγραφές οι οποίες προβλέπονται. Κατά τα άλλα ασχοληθήκαμε επίσης με την προστασία των ακτών διότι επί του θέματος αυτού έχουμε ε, και εμείς μία ψηφοφορία για την προστασία των ακτών. Η Ισπανία που έχει πολύ τουρισμό ίσως έχει περιοχές οι οποίες κινδυνεύουν όσον αφορά την ποιότητα του περιβάλλοντος και είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει εδώ και να, το, και να υπαγρυπνούμε. Και επίσης συζητήσαμε για την γεωργία και για την την εισαγωγή των, τον ε, ε, ε, με, τα αλλαγμένων οργανισμών στην Ισπανία. Τέλος πάντων ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα επίσκεψη. Πήγαμε και σε έναν σταθμό παρακολουθήσεως της φύσεως διότι θέλαμε να δούμε πώς γίνεται η παρακολούθηση των δασών στην Ισπανία και αυτό το οποίο είδαμε εκεί ήταν πραγματικά πολύ εντυπωσιακό ολίγης ε, αυτά είχα να σας πω σαν ε, επικεφαλής αντιπροσωπείας των 7 ατόμων θα ήθελα να κάνω μία τελευταία παρατήρηση δηλαδή ε, όταν υπάρχουν αντιπροσωπείες συνήθως είμαστε πολύ αυθόρμητοι και η κατάσταση είναι χαοτική και στο τέλος η αντιπροσωπεία δεν ήταν αντιπροσωπεία αλλά απλούστατα είχαν να απομείνει δύο από τα 7 μέλη και η γραμματεία θα πρέπει να ρωτάει εκ προημίου ποιος θα μείνει μέχρι πότε διότι δεν είναι ωραίο για αυτούς οι οποίοι μας φιλοξενούν να πηγαίνει μια αντιπροσωπεία η οποία σιγά σιγά εξατμίμεζεται και ε, πρέπει να σας πω ότι αυτό δεν είναι πολύ ευγενικό έναντι αυτών οι οποίοι μας υπεδέχθησαν. Αυτά είχα να σας πω σαν αφορά την εισαγωγή. Δεν ξέρω αν η Κάριν Καν θέλει να πει κάτι για την προστασία των δασών γιατί ήταν μία από τις δύο τελευταίες εναπομείνασες. Ε, αν όχι, ε, απλώς ε, σημειώνουμε τι εργασία έγινε, τι ε, ε, ε, τι προβλήματα υπάρχουν στη χώρα αυτή η οποία είναι μεγάλη μεν και έχει την προεδρία αυτή τη στιγμή πλην όμως δεν είναι όλα τέλεια και τέλος υπάρχει η έκθεση την οποία εγώ έχω αναλαβεί για τις αρμοδιότητες εφαρμογής την οποία θα ψηφίσουμε τώρα η τροπολογία 15 με split vote για το πρώτο μέρος. Ποιος είναι υπέρ του πρώτου αυτού μέρους. Ποιος είναι κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Μετά τροπολογία 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 19. 19. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 20 υπέρ ε, κατά αποχές απορρίπτεται. 21 υπέρ κατά αποχές εγώ το κάνω αυτό μετά. Split vote, ist für den split. 22 σε χωριστή ψηφοφορία ποιος είναι υπέρ του πρώτου μέρους κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο μέρος υπέρ. Λοιπόν, το δεύτερο μέρος καταπίπτει εφόσον το πρώτο μέρος απερίφθη με ειδοποιή γραμματεία και προχωράμε στην τροπολογία 23. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 27 ε, split, ε, χωριστή ψηφοφορία ε, σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος ποιος είναι υπέρ. Λοιπόν, μου λέγεται ότι το πρώτο μέρος καταπίπτει διότι έχουμε εγκρίνει την τροπολογία 24. αλλά έχει νόημα να ψηφίσουμε το δεύτερο μέρος. Οπότε ψηφίζουμε το δεύτερο μέρος της τροπολογίας 27 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 28 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 34 κατά Έλεγχο, ηλεκτρονικός έλεγχος ηλεκτρονική ψηφοφορία τελειώνει λοιπόν 24 υπέρ 28 κατά απορρίπτεται τροπολογία 7 υπέρ 7 ε, και 35 που είναι ταυτόσημες, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται να ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την, ε, τις τροπολογίες 7 και 35 λίγη απερίφθη 36 και 37 επίσης είναι ταυτόσιμες με μία προφορική τροπολογία. Ποιος είναι η υπέρ των τροπολογιών 36 και 37. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 38 υπέρ. καταπίπτει διότι ε, ε, απο, ε, αποδεχθήκαμε την 36 και 37. Τώρα ερχόμαστε λιμώντας το 8 καταπίπτει, το 1 απεσύρθη, τροπολογία 9, η οποία επίσης καταπίπτει. Η 10 όμως ισχύει. Μπορούμε λοιπόν να ψηφίσουμε το πρώτο μέρος της τροπολογίας 10. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο μέρος καταπίπτει. Και το τρίτο μέρος καταπίπτει επίσης. Τελευταία σελίδα. Τροπολογία 11. Καταπίπτει επίσης. 12. Ποιος είναι υπέρ της τροπολογίας 12. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το 13 καταργείται όπως και το 14. 4. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ερχόμαστε τώρα στην τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Το ΕΛΚ ε, έχει παραπάνω ψήφους. Ακόμη ένας περισσεύει από το ΕΛΚ. Τώρα όμως είμαστε εντάξει. Λοιπόν, 52 ε, ε, υπέρ και 5 αποχές, καμία αρνητική ψήφος ως εκ τούτου εγκρίνεται ε, αυτό το θέμα και σας ευχαριστώ ε, για την ψηφοφορία και προχωρούμε τώρα στο επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη ε, πρόταση για μια οδηγία του Συμβουλίου για τη χρήση ορισμένων επικινδύνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Έχετε μια σειρά από συμβαστικές τροπολογίες ενώπιόν σας που κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη, την ε, ψηφοφορία και καλώς εχόντων των πραγμάτων συνοψίζουν και ενοποιούν τροπολογίες πολλών μελών. Περνάμε λοιπόν στην ε, ψηφοφορία. Ενοποιημένη τροπολογία 1. Ψήφι υπέρ. Συμβαστική 1 λοιπόν. Υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβιβαστική τροπολογία υπαριθμών 2. Υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 3. Συμβαστική. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Ενοποιημένη τροπολογία 7. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ενοποιημένη τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος ηλεκτρονικός. Για την 4. Πέρας. Ψηφοφορίας. με μικρή, με μικρή πλειοψηφία απορρίπτεται. 29-27 απορρίφθηκε. Ενοποιημένη τροπολογία 5 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Είναι, είναι σαφές αν θέλετε μπορούμε να ελέγξουμε παρόλα αυτά για την 5. Κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο. Πέρας ψηφοφορίας. 33-23 ενεκρίθη λοιπόν, όπως φαινόταν και από πριν. Τροπολογία συμβασμού 6 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Άρθρο 1, τροπολογία 13 του εισηγητή ψήφι υπέρ κατά δεκτή Πάμε στη μέση της επόμενης σελίδας, στην 112, Sonic. Υπέρ της 112. Κατά αποχές δεκτή. Πάμε στη σελίδα 5. 1.44 του Chris Davis. Ψήφι υπέρ της 144. Κατά. Αποχές δεκτή. Επόμενη σελίδα, 145, πάλι Davis με προφορική τροποποίηση από τους πράσινους. Κύριε Σόνικ, είσαστε κατά ενίσταστε. Ωραία, οπότε μπορούμε να ψηφίσουμε μόνο το κείμενο ως είχε, βάσει του κανονισμού μας. Δεν μπορούμε να ψηφίσουμε την προφορική τροπολογία και εδώ υπάρχει αίτηση ψηφοφορίας κατά τμήματα σε τρία τμήματα συγκεκριμένα. Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα της 145 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Δεύτερο τμήμα ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα υπέρ. κατά αποχές απορρίπτεται και αυτό. Περνάμε στην επόμενη σελίδα. Τροπολογία Davis 152. Ψήφι κατά. Αποχές δεκτή. 19 της συγγήτριας. Ψήφι υπέρ κατά, αποχές, δεκτή. 20 συζυγήτριας υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 21 συζυγήτριας υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 22 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 156 υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. 23 υπέρ κατά άποχες δεκτή. 157-158 υπέρ κατά αποχές δεκτές. 25 συζυγήτριες υπέρ κατά άποχες εγκρίθηκε. Περνάμε στη σελίδα 9. 179 δεύτερο τμήμα της εισηγητρίας. Ψήφι υπέρ της 179 δεύτερο τμήμα. Ευχαριστώ. Κατά. Έλεγχος ηλεκτρονικός για την 179 τμήμα 2. Άρχεται η ψηφοφορία. Ένας από τους σοσιαλιστές περισσεύει. Εντάξει, ωραία τώρα είναι εντάξει. Πέρασε ψηφοφορίες. 25 υπέρ, 31 κατά, απορρίπτεται επομένω. Πάμε στην 183 και 317 που είναι με την 183. ψήφι υπέρ αυτών των δύο τροπολογιών. Κατά. Αποχές. <clears throat> Απορρίπτονται. Αυτοί που κατέθεσαν την τροπολογία την καταψηφίζουν τη δική του τροπολογία και αυτό είναι πρωτότυπο 190 ψήφι υπέρ. Σελίδα 10 είναι αυτό. Στη μέση της σελίδας 190 Chris Davis κατά αποχές απορρίπτεται. 191 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 192 υπέρ δεν, δεν πρέπει να ψηφιστεί εδώ λέει η γραμματεία η τροπολογία αυτή να μην ψηφιστεί εδώ. Ε, θα ψηφιστεί αργότερα μαζί με άλλες τροπολογίες. Πάμε στην 193. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. εκπίπτουν πολλές τροπολογίες, προχωρούμε, προχωρούμε, δεν ξέρω αν φτάνουμε μέχρι το τέλος κιόλας. Κάνουμε ένα μεγάλο άλμα και πάμε στη σελίδα 22, λέει ο πρόεδρος. Και συγκεκριμένοτερα την τροπολογία 50 της εισηγήτριας. 50 της εισηγήτριας. Ψήφι υπέρ. Σελίδα 22, τροπολογία 50 λοιπόν. Ψήφι υπέρ. <clears throat> Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ελπίζω να έχετε όλη την ίδια αριθμή σελίδα όπως και εγώ. Αλλιώς... Εντάξει. Εγώ βλέπω 22 και μετά 23. 151 λέει ο πρόεδρο τη εισηγήτριας υπέρ. Κατά <clears throat> απόχέ δεκτή. 2.74 Βέστλοντ. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχέ Απορρίπτεται. 52 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 53 της εισηγήτριας υπέρ κατά αποχές δεκτή. 54 της εισηγήτριας υπέρ κατά αποχές <clears throat> δεκτή. 2.75 βέστρον. υπέρ κατά αποχές δεκτή. 2.77 υπέρ κατά Έλεγχος ηλεκτρονικός για την 277. Τέλος πληροφορίας. Πολύ μικρή πλειοψηφία, 29-28 εγκρίνεται παρόλα αυτά. Άμα βγαίνετε από την αίθουσα, πληρώνετε αυτό. 2,76 Βέσλουντ. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 55 <clears throat> της εισηγήτριας. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 2,78, 2,79, 2,80 είναι ταυτόσιμες και οι τρεις. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτές. 56 έχει αποσυρθεί. 281 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 57 της εισηγήτριας υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 282 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 58 τη εισηγήτριας υπέρ, κατά, <clears throat> αποχές δεκτή. 283, 284, 285 ταυτόσιμες ψήφοι υπέρ, κατά, αποχές δεκτές. 286-287 ψήφοι υπέρ. Ψηφίζονται μαζί αυτές. Κατά, άποχες, δεκτές. 61 τη υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 62, υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 2.88 Ντέβις, υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 63 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 64 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 2.89 ψήφι υπέρ κατά έλεγχος. 2.89 Άρχιντη ψηφοφορία. Πέρασε ψηφοφορίας. Δεκτή 32-26. 2,92 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Διακόσια 291 ψήφι υπέρ, κατά, άποχες, δεκτή.

ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 67 της εισηγήτριας. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράτημα 3, τροπολογία 306 Σόνιξ στη σελίδα 25, που ταυτίζεται με την 307-308. Ψήφι υπέρ των τριών αυτών τροπολογιών. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. Τροπολογία 70 Τη εισηγήτριας, το πρώτο τμήμα δεν χρειάζεται να ψηφιστεί ήδη. Ψηφίζουμε το δεύτερο, τρίτο, τέταρτο αλλά και πέμπτο τμήμα. Δεύτερο τμήμα πρώτα, της 70. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. Έλεγχος μάλιστα. Άρχεται η ψηφοφορία για το δεύτερο τμήμα. Πέρας ψηφοφορίας. Το ΕΛΚ έχει ένα παραπάνω που ψηφίζει. Εντάξει, αποσύρθηκε μία κάρτα. 30 με 28 εγκρίνεται το δεύτερο τμήμα. Τρίτο τμήμα. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ίδια πλειοψηφία πιστεύω. Θέλετε να ελέγξουμε και πάλι. Άρχεται ηλεκτρονικό έλεγχο για το τρίτο τμήμα. Εγώ πιστεύω θα είναι ακριβώς η ίδια πλειοψηφία. Τέλος τη προφορίας. Σχεδόν η ίδια πλειοψηφία. 29-28 λέει ο πρόεδρος. Κάποιος ξέχασε να ψηφίσει. Δεκτό το τρίτο τμήμα λοιπόν. Τέταρτο τμήμα. Τέταρτο τμήμα ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Πάλι ηλεκτρονικός έλεγχος για το τέταρτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Λίγο μεγαλύτερη διαφορά, 29-27 δεκτό, πέμπτο τμήμα τώρα. Ψήφι υπέρ του πέμπτου τμήματος, κατά. Αυτό είναι φανερό. Απορρίπτεται σαφώς. «310 πρώτο τμήμα. Ψήφι υπέρ». Κατά. Έλεγχος. Για το 310 πρώτο τμήμα. μικρη Μικρή διαφορά, 29-28, εγκρίνεται. 311, ψήφι υπέρ. Κατά. Έλεγχος. 311. περας ψηφοφορία. ψηφοφορίας. 30-28 εγκρίνεται. 309 τμήμα 1 ψήφι υπέρ. Κατά. Δεκτό. Δεκτή η τροπολογία. Έλεγχος. Έλεγχος για το, την 309 τμήμα 1. Πέρας. Άξιζε τον κόπο. 29-29 απορρίπτεται λόγω οψηφίας. απορρίπτεται λοιπόν. 314. πρώτο τμήμα. Που ταυτίζεται με την 313 πρώτο τμήμα. Αλλά και με την 315 πρώτο τμήμα. Μοιάζουν να είναι ακριβώς οι ίδιες. Ψηφίζουμε αυτές τις τρεις τροπολογίες, πρώτο τμήμα, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. «71 της εισηγήτριας και αυτή περιλαμβανόταν στις ε, ταυτόσιμες τροπολογίες. 314 δεύτερο τμήμα που ταυτίζεται με την 71 δεύτερο τμήμα. Κοινή ψηφοφορία λοιπόν ψηφίπερ. Κατά αποχές απορρίπτονται. 313 τμήμα 2 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 3.14 τρίτο τμήμα και 71 τρίτο τμήμα ψήφι υπέρ των δύο τροπολογιών <clears throat> κατά αποχές απορρίπτονται. 3.13 τρίτο τμήμα ψήφι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 314 τέταρτο τμήμα, 71 <clears throat> τέταρτο τμήμα, 313 επίσης τέταρτο τμήμα, ψήφι υπέρ αυτών των τροπολογιών. Κατά αποχές απορρίπτονται. 314 πέμπτο τμήμα, 71 πέμπτο τμήμα, 313 πέμπτο τμήμα, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτονται. 314 έκτο τμήμα, 70, ναι, αυτή μονάχα είναι η ψήφι υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτονται. 71 έκτο τμήμα, 313 έκτο τμήμα, ψήφι υπέρ, κατά άποχες απορρίπτονται. 313 έβδομο τμήμα ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. «315, δεύτερο τμήμα, Φανμπρέμπτ Μέρκες, ψήφι υπέρ» κατά αποχές απορρίπτεται. Προχωρούμε. 319 Γκέλιν και 320 Ντέβις που είναι ταυτόσιμες υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Έλεγχος βεβαίως. 319-320. 32 προς 25 γίνονται, γίνεται δεκτή. Γίνονται δεκτές μάλλον. 321 και 322 που είναι ταυτόσιμες. Ψήφι υπέρ. Κατά. Άποχες. Δεκτή. 323-324. Ταυτόσιμες. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές δεκτές. 325-326 ταυτόσιμες ψήφι υπέρ κατά αποχές δεκτές. 328-329 ταυτόσιμες ψήφι υπέρ κατά αποχές δεκτές. 327 ψηφι υπέρ κατά αποχές δεκτή. 3.30-3.31 ταυτοσιμες ψήφοι ψήφι υπέρ, κατά, αποχές δεκτές. 3.32-3.33 ταυτόσιμες ψήφοι υπέρ, κατά, αποχές δεκτές. 3.34 ε, ψήφοι υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. τροπολογία 75 της εισηγήτριας. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 76 και 339 ταυτίζονται ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. αιτιολογικές σκέψεις. 1. Εισηγήτριες υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 79. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Έλεγχος. Για το 79. Ένας σοσιαλιστής περισσεύει. Ε, Τζιλ πρέπει κάποιος να αποσυρθεί. 31-27 εγκρίνεται. Δύο της εισηγητρίας <clears throat> ψήφι υπέρ. Κατά αποχές δεκτό. 5. Πέντε ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. ογδόντα δύο ταυτόσιμες, ψήφι υπέρ. κατά αποχές δεκτά. 83 ψήφοι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 84 ψήφοι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. 85 καθώς και 86 ταυτόσιμες ψήφοι υπέρ. κατά αποχές δεκτό. Οχτώ της εισηγήτριας υπέρ κατά αποχές εγώ νομίζω ότι έχει εγκριθεί αλλά αν θέλετε κάνουμε έλεγχο ηλεκτρονικό για το 8 Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 31-27 εγκρίνεται. 89 με, χωρισ... με ψηφοφορία σε τμήματα. Πρώτο τμήμα ψήφι υπέρ. Κατά αποχές δεκτό. Δεύτερο τμήμα, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Αυτά ήτανε. Τελειώσαμε. Θαυμάσια. Θαυμάσια λέει ο πρόεδρος. Τελική ψηφοφορία για το σχέδιο εκθέσεως όπως τροποποιήθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ένας από το ΕΛΚ περισσεύει. Τώρα εντάξει. Πέρας ψηφοφορίας. 55-1 με δύο αποχές. Συντριπτική πλειοψηφία. Το νομοθετικό ψήφισμα. Πάλι ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. 53 υπέρ, καμ... καμία ψήφος κατά, μία αποχή. Συντριπτική πλειοψηφία. Συγχαίρω και πάλι την εισηγήτρια. Με μία πάρα πολύ σημαντική έκθεση. Είναι σημαντική για την ε, στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι της κλιματικής αλλαγής Έχουμε συμβάλει λοιπόν στη διαμόρφωση μιας i4 στρατηγικής στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Τώρα είναι πιο απλά τα πράγματα. Ερχόμαστε <clears throat> στο επόμενο θέμα. Η σύναψη του πρωτοκόλου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παρακτήων ζωνών της Μεσογείου στη Σύμβαση για την Προστασία του Θαλασσίου Περιβάλλοντος και των Παρακτήων Περιοχών της Μεσογείου. Μπορούμε να πούμε είτε ναι είτε όχι, ε, διότι υπάρχει μόνο μία ψηφοφορία. Ποιος είναι υπέρ αυτού του ψηφίσματος. Κατά αποχές ε, θα πρέπει να γίνει και ηλεκτρονικός έλεγχος. Ξεκινάει η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Λίγοι. 53 υπέρ, κανείς κατά, καμία αποχή, ομόφωνα α, υιοθετείται για την καλύτερη προστασία των ακτών στην Ευρώπη. Ε, τώρα ερχόμαστε στο επόμενο θέμα, πράσινη βίβλος της Επιτροπής για τη διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εισηγητής ο Χωσέ Μανουέλ Φερνάντες. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ερχόμαστε τώρα στην πρώτη συμβιβαστική. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2. Ποιος είναι υπέρ της συμβιβαστικής 2. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Μετά, ε, τροπολογία 54 Βαμπρέμπτ. Όχι. 58 ε, Μαγκίνες. Ποιος είναι υπέρ της τροπολογίας 58. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 79 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 57 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Λίγοι. Ήτανε τσίμα τσίμα με μία ψήφο απερίφθη. 61 υπέρ. Κατά. Ε, δεν βλέπω ότι γίνεται. Ας ελέγξουμε και την 61. Παρακαλώ, σηκώνετε καλά τα χέρια σας, διαφορετικά δεν βλέπω. Ξεκινάει ηλεκτρονικός έλεγχος. Λίγοι. 29 υπέρ, 23 κατά, άρα εγκρίνεται. 60 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 59 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ταυτόσιμες οι 65 και 66 αλλά βλέπω ότι όλες τις τροπολογίες της παραγράφου 4 όλες έχουν αποσυρθεί λόγω της πρώτης συμβιβαστική. και προχωρούμε στην 67 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 68 με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 69 υπέρ κατά απορρίπτεται 70 χωριστή ψηφοφορία πρώτο μέρος ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 74 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 75 κατά αποχές απορρίπτεται 76 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 77 κατά αποχές απορρίπτεται 81 Παναγιώτοφ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 78 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τώρα ερχόμαστε στην τρίτη τροπολογία της Επιτροπής Γεωργίας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4 ε, άγκρι υπέρ κατά Αποχέ, εγκρίνεται άγκρι 5 υπέρ κατά απόχέ. απορρίπτεται άγκρι 6 υπέρ κατά απόχέ, εγκρίνεται άγκρι 7 υπέρ κατά Αποχέ εγκρίνεται άγκρι 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 υπέρ άγκρι 9 Απο, ε, ε, ε, αποδεκτή το άγκρι 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται άγκρι 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται για την άγκρι 12 όχι, όχι, το, την καλύψαμε. Άγκρι 13, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Άγκρι 14, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Άγκρι 15, υπέρ. Κατά. αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την άγκρη 15. Λίγοι. 33 υπέρ 25 κατά εγκρίνεται. Ε, Άγκρι 16 χωριστή ψηφοφορία σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται άγκρι 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται άγκρι 18 χωριστή ψηφοφορία πρώτο μέρος ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άγκρι 19 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Άγκρι 20 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Άγκρι 21 υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονικός έλεγχος της Άγκρι 21. Λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 24 υπέρ, 31 κατά. Ήτρε 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα έλεγα ότι απερίφθη, αλλά κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο για την Ήτρε 1. Το ΕΛΚ έχει έναν παραπάνω, οπότε δεν μας απασχολεί. Στο σχόλιο το οποίο δεν ακούστηκε γιατί τα χωρίς μικρόφωνο. 26 υπέρ, 31 κατά, απερίφθη. Ήτρε 2. Ε, κατά. με πλειοψηφία περίφθη. Ήτρε 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ήτρε 4 χωριστή ψηφοφορία πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ήτρε 5 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ήτρε 8 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ήτρε 9 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 10 Ήτρε υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ήτρε 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ήτρε 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ήτρε 13 με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ήτρε 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ήτρε 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ήτρε 17 με χωριστή ψηφοφορία, πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ήτρε 18 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ήτρε 19 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. εκτιμώντας. 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 5. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 9 υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 13 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 14. Με προφορική τροπολογία και χωριστή ψηφοφορία. Πρώτα η προφορική, ψηφοφορία, η προφορική τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Χωριστή ψηφοφορία πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για το δεύτερο τμήμα μάλιστα. Ε, ένα σοσιαλιστής και ένα σέλκ παραπάνω. ακόμη περισσεύει κάποιος σοσιαλιστής. Τώρα όμως είμαστε εντάξει. Απερίφθη. 32 κατά και 25 υπέρ. Θα μπορούσε να έχει περάσει αλλά δεν πέρασε. 15. Ποιος είναι υπέρ της τροπολογίας 15. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 16. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα ερχόμαστε στη συμβαστική 4. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 21. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 23 υπέρ κατά Βλέπω ότι στην επόμενη σελίδα υπάρχει ε, μία χωριστή ψηφοφορία για την τροπολογία 23 πρώτο μέρος. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 24 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 32, τροπολογία 32, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ελέγχουμε την 32. Από το ΕΛΚ πάλι περισσεύει κάποιος. Κάποιος πρέπει να βγάλει την κάρτα του. Εντάξει, τώρα είμαστε εντάξει. Λίγη ψηφοφορία. Ε, με μικρή πλειοψηφία, 29 υπέρ, 28 κατά και μία αποχή. Μετά, το εκτιμώντας ε, ε κάπα, τροπολογία προφορική Ρώση. Ε, υπάρχει αντίρρηση στην ε, προφορική τροπολογία, αλλά δεν μπορούμε να την ψηφίσουμε. Και ψηφίζουμε το αρχικό κείμενο. Ποιος είναι υπέρ του αρχικού κειμένου. Ποιος είναι κατά. Απορρίπτεται. Επόμενο, τροπολογία 33. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 38 και 39 ταυτόσημες υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 37. Ποιος είναι υπέρ της ορπολογίας 37. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 34. τέσσερα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία Ρώση. Αν δεν υπάρχει αντίρρηση την ψηφίζουμε. Ποιος είναι υπέρ της προφορικής τροπολογίας Ρώση. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 40 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 41 με προφορική τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 42. Βαν Μπρέμπτ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ε, ηλεκτρονικός έλεγχος τροπολογία 43 Λίγη ψηφοφορία πάλι ε, ε, πολύ τσιμα τσιμα αλλά πέρασε 29 υπέρ 28 ε, κατά 44 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 45 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και φτάνουμε στην τελική ψηφοφορία η οποία θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά. Ξεκινά. Δύο ΕΛΚ περισσεύουν. Νο, ακόμη ένας περισσεύει. Μία κάρτα πρέπει να αφαιρεθεί. Τώρα είμαστε εντάξει. Λίγη ψηφοφορία, 55 υπέρ, 3 κατά, καμία α, αποχή και συγχαίρω τον εισηγητή Χωσέ Μανουέλ Φερνάντες. Σημείο υπαριθμών 9. δίκαια εισοδήματα για του αγρότε και βελτίωση της λειτουργία τη αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων στην Ευρώπη. Η εισηγήτρια είναι η Εστέρ Εράν Γκαρθία. Ψηφίζουμε τροπολογία υπαριθμών 1. ποιο είναι υπέρ. Κατά. Άποχε. Δεκτή. 2 υπέρ. Κατά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 κατά αποχές εγκρίνεται. 11 με χωριστή ψηφοφορία σε τμήματα. Πρώτο τμήμα, ψήφι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κα, υπέρ. Δεύτερο τμήμα, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 12, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 13 υπέρ κατά αποχές δεκτό 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 18 σε τμήματα, πρώτο τμήμα, ψήφι υπέρ, κατά, έλεγχος για το πρώτο τμήμα της 18. Πέρας. Ενεκρίθη σαφώς. Δεύτερο τμήμα, ψήφι υπέρ κατά αποχές δεκτό. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 54-2 καμία αποχή εγκρίνεται λοιπόν Συγχαρητήρια στην εισηγητρία την Εστέρ Εράν Γκαρσία. Ευχαριστούμε για την εργασία σα για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Περνάμε στην ανάπτυξη του δημιουργού δυναμικού συγγνώμη, δημιουργίας θέσεων στα πλαίσια μιας νέας βιώσιμης οικονομίας. Η συγγήτρια κυρία Ροβάνα Πλάμπ Συγχαρητήρια για την παρθενική σας ε, έκθεση, κυρία Πλάμπ. Τροπολογία 1. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 2. <clears throat> με προφορική τροποποίηση υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή υπερθυμών 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 8 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές <clears throat> απορρίπτεται. 9 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 10 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 12 <clears throat> με προφορική τροποποίηση υπέρ κατά αποχές δεκτή. 13 με προφορική τροποποίηση ψήφι υπέρ κατά αποχές δεκτή. 14 υπέρ κατά Αποχές απορρίπτεται. 15 ψήφι υπέρ. Κατά. Δεκτή. 16 με τρο... προφορική τροποποίηση ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 17 με προφορική τροποποίηση και χωριστή ψηφοφορία. 16 θέλετε έλεγχο. Έλεγχος για τη 16. Εντάξει. Πέρας ψηφοφορίας. Α, απορρίπτεται. 25 υπέρ, 30 κατά. Απερίφθη η 16. 17. Με προφορική τροποποίηση και χωριστά και δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές δεκτό. Αυτό ήταν μάλλον την προφορική τροποποίηση. Ε, την ψηφοφορία, πρώτο τμήμα. Κατά. Αποχές, δεκτό. Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά. Άποχες, έλεγχος για το δεύτερο τμήμα, της 17. Πέρας. 30-25 εγκρίνεται. 18. με Ρίτ Μακίνες ψηφί υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 19. Χωριστή ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ κατά αποχές δεκτό. 20 ψήφι κατά αποχές δεκτή. 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Άρχεται ψηφοφορία. πέρα περας προφοριες προφορίας. 53-1 με μία αποχή μονάχα. Συγχαρητήρια στην κυρία Ροβάνα Πλόμπ. Και έχουμε εργαστεί πάρα πολύ ωραία. Εξαιρετικά έχει τελειώσει η ημερησία διάταξη του της πρωίας και έχετε δύο ώρες για να κάνετε κάτι πιο επωφελές. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία σας. Τρεις η ώρα συνεχίζουμε. Ah,